την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλουν τις λειτουργίες των whistleblowers. Εξ ονόματος του Συμβουλίου και της ε, νέας Σλοβακικής Προεδρίας ε, το λόγο έχει ο κύριος Κόρτσοκ. Uh, Κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι για πρώτη φορά εμφανίζομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τότε που ανέλαβε την Προεδρία η Σλοβακία. Είναι η πρώτη μας άλλωστε Προεδρία, ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ευθύ εξ αρχή να πω ότι είμαστε πεπισμένοι ότι εδώ εκπροσωπώντας το Συμβούλιο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε ξεκάθαρες προτεραιότητες. Βασίζομαι λοιπόν σε εσά ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε απτά αποτελέσματα. Περισσότερο από ποτέ πρέπει να έχουμε απτά αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συζητήσουμε το ζήτημα της προστασίας των υπαλλήλων που καταγγέλνουν τις λειτουργίες των πληροφοριοδοτών Ξέρετε ότι έχουμε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια που κατέδειξαν τον ρόλο που διδραματίζουν οι καταγγέλτες σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Όταν προστατεύει κανείς το κοινό δημόσιο συμφέρον, προφοριοδότες διδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Καταδεικνύουν παρατυπίες και κινδύνους, θα έλεγα, στα πλαίσια της κοινωνίας μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να καταγγέλουν και να προδοποιούν κάθε φορά χωρίς να χρειάζεται να καταβάλουν ένα σημαντικό τίμημα την ίδια τη φήμη τους, τη ζωή τους, τη δουλειά τους. Η ε, προστασία λοιπόν των ανθρώπων αυτών, των πληροφοριδιωτών, αποτελεί αντικείμενο διαφόρων διεθνών μέσων επί του παρόντος. Για παράδειγμα έχουμε τις κατευθυντήρες γραμμές του ΟΣΑ του 2012, Παράλληλα, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει μια σύσταση ήδη από το 2014 όπου ζητά από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλνουν τις λειτουργίες. Στο επίπεδο τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διάφορα νομοθετήματα τα οποία περιέχουν διατάξεις για την προστασία των ανθρώπων αυτών, όπως για παράδειγμα η προστασία των δημοσιογράφων που καταγγέλουν παρατυπίες, ζήτημα το οποίο συζητήσαμε στα πλαίσια της οδηγίας για το εμπορικό απόρριτο πέρυσι. Προβλέπεται εδώ πέρα προστασία λοιπόν για τους καταγγέλτες κάθε φορά που αποκαλύπτουν παρατυπίες ή παράνομες δραστηριότητες αρκεί βέβαια να έχουν δράσει προς το κοινό καλό για το δημόσιο συμφέρον. Επίσης Παρόμοιε διατάξει έχουμε σε διάφορε οδηγίε ή κανονισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίω όσον αφορά τι χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε. Διατάξει επίση υπάρχουν και σε επίπεδο εθνική νομοθεσία, ιδίω στα πλαίσια των συστάσεων του Συμβουλίου τη Ευρώπη που ανέφερα πριν από λίγο. Όσον αφορά τώρα μια πιο οριζόντια νομοθεσία που θα μπορούσαμε να είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο και καταγράφω πάντως την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελτών μέχρι τα τέλη του Ιουνίου του 2016. Προσβλέπω λοιπόν να ακούσω την παρέμβαση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα αυτό. Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα συζητήσει εις βάθος το ζήτημα. Πάντως γενικότερα έχει προσεγγίσει το ζήτημα αυτό όσον αφορά τις πολιτικές που θα μπορούσαμε να είχαμε στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Αξιότιμα μέλη, Ολοκληρώνοντας, θα έλεγα ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του το Συμβούλιο είναι έτοιμο να εξετάσει μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα αναγκαία ευρωπαϊκά μέτρα για την προστασία των υπαλλήλων που καταγγέλουν λειτουργίε. Ήδη από χθε ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για τα επόμενα μέσα, τα μελλοντικά μέσα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στην καταπολέμηση τη φοραποφυγής και φοροδιαφυγής. Και αυτό συνδέεται με τους καταγγέλτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρω ότι θα εξετάσει την δυνατότητα μιας οριζόντιας νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας όμως υπόψη και την αρχή της επικουρικότητας. Σας ευχαριστώ. Εξ της Επιτροπής, το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος κ. Κατάινεν. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να συζητήσω μαζί σας την προστασία των καταγγελόντων μετά από τη συζήτηση που έγινε εδώ τέσσερις μήνες πριν. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ορίσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο προστασίας τους και να υπάρχει και λογοδοσία. Θα πρέπει να προστατευτούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δυσλειτουργίες και παρατυπίες καθώς και εγκληματικές δραστηριότητες. Γι' αυτό η Επιτροπή τάσεται υπέρ της προστασίας των καταγγελόντων. Και αυτό μέσα στα πλαίσια και της τομεακής νομοθεσίας μας και της νομοθεσίας της 6 Δεκεμβρίου 2012. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ορίσουν αξιόπιστους ε, μηχανισμούς έτσι ώστε να καταγγέλλονται οι παρατυπίες ε, στον κρατικό μηχανισμό, ιδιαίτερα σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος. Επίσης έχουν τεθεί οι υπό εφαρμογή οι διαδικασίες αυτές έτσι ώστε να μην γίνονται παραβιάσεις αυτών των κανόνων. Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα γραφεία ορκωτών ε, ε, λογιστών και τα γραφεία νομικών συμβουλών. Και επίσης όσον αφορά την ε, μεταφορά χρεογράφων τα έγγραφα του Παναμά τόνισαν τη σημασία της εφαρμογής αυτής της ε, ρήτρα έτσι ώστε να ε, γίνονται έρευνες για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή γι' αυτό. Συντάξαμε μία ανακοίνωση όπου γίνεται λόγος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή και τις παράνομες χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. Επίσης προβάλλουμε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών έτσι ώστε να προβάλλουμε την προστασία σε εθνικό επίπεδο. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να μιλήσω για την διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης μέσα στα πλαίσια του ε, πλουραλισμού, στα πλαίσια του δεύτερου συμποσίου που θα λάβει υπόψη, που θα λάβει, συγγνώμη, χώρα κατά τα τέλη Οκτωβρίου αρχές Δεκεμβρίου του 2016 σε σχέση με τα δικαιώματα των καταγγελόντων και αυτό αφορά και την πίεση σε δημοσιογραφικές πηγές και αυτό φυσικά αφορά και τους καταγγέλλοντες. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε και ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει πολλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εκεί όπου, που, όπου έχουμε αρμοδιότητα, για να ενισχύσουμε τη θέση των καταγγελόντων. Θα πρέπει να τονίσουμε το, ε, τα οριζόντια και κάθετα επίπεδα εφαρμογής της νομοθεσίας μέσα στα πλαίσια της ε, αλληλεγγύης. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας στα θέματα αυτά και προσβλέπουμε θετική συνεργασία. Περνούμε στον κύκλο των ομιλητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για την ομάδα του Λαϊκού Κόμματος. Το λόγο έχει η κυρία Πιτέρα για δύο λεπτά. Dziękuję, panie przewodniczący. Konwencja na... Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σύμβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς που έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνει το άρθρο 33 για την προστασία των καταγγελόντων και καλεί τα, τα μέρη ε, στα νομικά του συστήματα ε, να εγγυώνται τα δικαιώματα και την ασφάλεια αυτών των ατόμων που καταγγέλνουν παρατυπίες. Επίσης, η αντίστοιχη σύμβαση περί του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, έχει το άρθρο 9 που υποχρεώνει τα συμβολόμενα μέρη να προστατεύουν τους καταγγέλλοντες. Και οι δύο αυτές συμβάσεις αναφέρουν ότι αυτοί οι οποίοι δρούν καλή την πίστη θα πρέπει να προστατεύονται. Και οι καταγγέλλοντες πρέπει να προστατεύονται επειδή ακριβώς γνωρίζουν την εσωτερική λειτουργία κάποιου θεσμού και είναι αυτοί που πιο γρήγορα μπορούν να ε, καταγγείλουν και να εκθέσουν αυτούς που παρατυπούν. Η δράση τους έχει άμεση σχέση με την αποκάλυψη παρατυπιών και ε, πρέπει να προστατεύονται υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δρούν καλή την πίστη και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Τον Ιούλιο του 2011 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε κάλεσε μάλλον τα κράτη-μέλη να προστατεύουν τους καταγγέλλοντες παρατυπίες μόνο όταν οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από αυτούς ε, είναι σαφώς και καταφανώς υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Το Νοέμβριο του 2012 το ίδιο ε, δικαστήριο ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να περιορίζουν ή να μειώνουν την δυνατότητα καταγγελών και δημοσιογράφων να ε, εκθέτουν και να καταγγέλουν παράνομες παράτιμες πράξεις υπό την προπόθεση ότι αυτό γίνεται υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και καλή την πίστη. Ένα δίκαιο σύστημα προστασίας λοιπόν είναι απολύτως απαραίτητο αν θέλουμε να μειώσουμε τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Ρενιέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Πίτροπε, κύριε Κατάινεν. Ε, θα ήθελα άμεσα να σας πω αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Χρειαζόμαστε μια οριζόντια οδηγία, μια γενική οδηγία η οποία να προστατεύει εν γέρι τους καταγγέλλοντας και όχι μόνο ε, σε τομακό επίπεδο. Αυτό δεν είναι θέμα, ε, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλεσης, όχι της νομικής βάσης, γιατί υπάρχει μια νομική βάση. Εάν ε, η Επιτροπή προτίθεται να πάει παραπέρα, είναι κάτι τέτοιο απολύτως εφικτό. Γι' αυτό ε, θεωρώ ότι αποτελεί ένα θετικό νεύμα ότι μπορούμε να, μπορεί να γίνει κάτι και νομίζω ότι η συζήτηση αυτή γίνεται σε σωστό χρονικό ε, σημείο γιατί εάν δούμε την απόφαση η οποία ελήφθη την περασμένη εβδομάδα ε, η οποία είναι επονίδιστη για την Ευρώπη γιατί άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά δρούν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος απολύονται. Άρα λοιπόν και κάποιος ο οποίος έχει ε, κερδίσει ένα βραβείο για, το, για τα επιτεύγματά του τελικά ε, τιμωρείται. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οριζόντια οδηγία, όχι μια η οποία λειτουργεί σε τομεακό ε, επίπεδο. Εάν δούμε τι γίνεται με τα Lux Leaks, όταν το διακύβευμα είναι αυτών των διαστάσεων, ε, θα πρέπει ακριβώς να μπορούμε να υπολογίσουμε σε αυτή την ε, συνεργασία και στην ε, βοήθεια τη συνεισφορά των καταγγελόντων. Η Επιτροπή έχει φτάσει να το αναγνωρίσει αυτό και είμαι βέβαιο ότι θα την υποστηρίξει και το Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε κυρία Μακοβέη. Ευχαριστώ. Σίγουρα θα, θέλουμε να, θα θέλαμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και στα εθνικά ως προς τις παρανομίες και παρατυπίες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε θαραλέους ανθρώπους και αξιοπρεπείς που να εργάζονται στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών αρχών. Πιστεύω ότι προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον έτσι ώστε να σταματήσουν τις παρατυπίες και τις παρανομίες σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε και δεν υπάρχει αντίστοιχη πολιτική προστασίας. Διαφορετικά θα χάσουν τη θέση εργασίας τους. Εγώ παρακολουθώ ανθρώπους που δουλεύουν σε διάφορα όργανα οι οποίοι μου, μου μίλησαν για παρατυπίες αλλά φοβούνται να τις καταγγείλουν. Πρέπει να τους, να τους προστατεύσουν. Κύριε Παγκαθουρτούντουα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Όταν ακούω για να μιλάμε για αυτές τις οδηγίες, τους κανονισμούς και όλα τα σχετικά, ε, σκέφτομαι σαν να βρισκόμαι στο, στην ε, χώρα της συναλήξης των θαμάτων, που κυνηγάμε ε, το καπέλο που μας ξεδιφεύγει συνεχώς, σαν να είμαστε ο λαγός δηλαδή. Γιατί σαν να μας διαφεύγει. Η οδηγία του 2014 αναθεώρησε ε, την συμφωνία που είχαμε καταλήξει, στην οποία είχαμε καταλήξει με πολλές χώρες, εκτός από τον Παναμά όμως το, ε, όλα, όλα καλύφθηκαν μετά από μια ανώνυμη καταγγελία. Ε, αλλά ε, σε άλλες περιπτώσεις ε, όσοι κατήγγυλαν επώνυμα είχαν πολλές φορές σημαντικές βλάθηκαν τα συμφέροντά τους σε μεγάλο βαθμό. Θα πρέπει να τους προστατεύσουμε. Τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Η ομάδα μου θεωρεί ότι οι καταγγέλλοντες ε, παίζουν ζωτικό ρόλο στην προστασία της δημοκρατίας υπέρ του γενικού συμφέροντος. Ε, τα Panama Papers ή τα διάφορα leaks ε, αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε τα νομικά μέσα που χρειάζονται για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και θα πρέπει να προστατεύουμε τους καταγγέλλοντες. Ο ε, καταγγέλθηκε, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλακή και σε πρόστιμο παρόλη στην προστασία που υποτίθεται υπάρχει. Ε, η ατιμορρησία είναι το χειρότερο στοιχείο το οποίο θα μπορούσαμε να εισάγουμε στα ε, όργανά μας και στους φορείς μας. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε με οριζόντια οδηγία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, η αριστερά ζήτησε μια τέτοια συζήτηση στο Λουξεμβούργο. Ο Ραφαέλ Αλέφ και ο Βάντε Τούρ ε, καταδικάστηκαν επειδή ενημέρωσαν την κοινή γνώμη για τα Λουξ ε, λίξ ε, και αυτό έγινε υπό την ευθύνη του παρόντος ε, Προέδρου της Επιτροπής του Ζαν Κλοντ Juncker. Η Apple και η Google πληρώνουν λιγότερο από 1% φόρων επί των κερδών τους και χρειαζόμαστε ε, και χάνουμε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως ε, χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για την οικοδόμηση σχολείων. Ε, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι ε, καταγγέλουν μια ποινικά κολάσιμη πράξη δεν θα έπρεπε να καταδικάζονται αλλά θα έπρεπε οι δράστες να τιμωρούνται. Ο Αντουάν ε, κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο των Πολιτών και το έργο του αξιολογήθηκε θετικά. Αυτό όμως που χρειάζονται οι ήρωες είναι προστασία και όχι παχιά λόγια. Ο κύριος Γιούγκερ είπε ότι χρειάζεται μια προστασία των καταγγελών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο δεν έχει συμβεί μέχρι τίποτε. Παρακαλέσαμε τους ε, ε, σοσιαλδημοκράτες και το Λαϊκό Κόμμα να μην ψηφιστεί εν λόγω ειδηγία πριν εξασφαλιστεί η προστασία, επαρκώς η προστασία των καταγγελόντων αλλά δεν εισακουστήκαμε. Ο συνάδελφος De Jong ε, θα υποβάλει ε, μια έκθεση όσον αφορά την ε, προστασία των καταγγελόντων σε σχέση με τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ να υποστηρίξετε την εργασία του Ντένις, γιατί πραγματικά θα πρέπει να παρασχεθεί η προστασία αυτή, οτιδήποτε άλλο θα ήταν πονίδιστο. Ευχαριστώ κύριο Ντυρό. Κυρία Ντυρό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επιτρόπε που αναφέρατε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τους καταγγέλλοντες. Πέρα από τα λόγια όμως το σημαντικό είναι να περάσουμε στις πράξεις. Βρισκόμαστε σε ένα κόσμο παράξενο. Αυτοί οι οποίοι καταγγέλνουν τις παρατυπίες ε, καταδιώκονται και τιμώνονται από τη δικαιοσύνη. Ενώ τα άτομα τα οποία καταγγέλλονται τη βγάζουν καθαρή. Ένα αλόκοτο κόσμος όπου οι δημοσιογράφοι που πληροφορούν την κοινή γνώμη ε, απολύονται. Αυτοί όμως ε, οι οποίοι ε, καταγγέλλονται ε, δεν βαθαίνουν τίποτα. Ε, αυτή είναι η ελεύθερη πληροφόρηση δεν θα έπρεπε να προστατεύονται αυτά τα άτομα. Γιατί θα πρέπει να προστατεύονται, για τον εξή πολύ απλό λόγο. Γιατί είναι οι φύλακε, οι θεματοφύλακε του γενικού δημόσιου συμφέροντο. Ε, είναι οι θεματοφύλακε μια ανοιχτή και διάφανη δημοκρατία. Για λόγου περιβάλλοντο, για λόγου υγεία, για φορολογικού λόγου, για διαφθορά, οτιδήποτε και να καταγγέλλεται, χρειαζόμαστε αυτές τις, αυτούς τους ανθρώπους και πρέπει να τους προστατεύουμε, όχι να τους φυλακίζουμε και να τους διώκουμε. Θα ήταν τιμητικό για την Κομισιόν να σεβαστεί αυτό που έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε γρήγορα να υποβάλει ένα κείμενο, να πάρει δηλαδή την πρωτοβουλία η Κομισιόν, ε, να καλύψει τα κενά τι αδυναμίες που υπάρχουν. Γιατί δεν το κάνετε. Εμείς εκ μέρους των οικολόγων σας ζητούμε να υποβάλλετε ένα οριζόντιο ευρωπαϊκό κείμενο για υπέρ ε, του δημοσίου συμφέροντος προστασίας αυτών των ατόμων. Ευχαριστώ. Η κυρία Φεράρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα διονγκούμενα φαινόμενα ε, διαφόρων παράτυπων και παράνομων δραστηριοτήτων, της διαφθοράς, οι πολυεθνικές, οι οργανισμοί που συμπεριφέρονται παράνομα, υποθάλπουν, υποθάλπτουν συγγνώμη, τη δραστηριότητα και τη ζωή των πολιτών. Και αυτά είναι δόλια φαινόμενα που βλάπτουν την ε, κοινωνία. Οι κρατικές αρχές δεν τα καταφέρουν γιατί ορισμένα φαινόμενα είναι δύσκολο να αποκαλυφθούν. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους πολίτες έτσι ώστε να καταγγέλουν τις παράνομες δραστηριότητες αυτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εισαγάγει ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των καταγγελόντων. Μετά από το Lux Leaks βλέπουμε ότι δεν έχουμε πια χρόνο να χάσουμε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πρέτσελ δεν είναι παρόν. Έτσι φαίνεται. Η κυρία Λεγκρίπ λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπό την ιδιότητά μου ως εισηγήτρια της, ε, για την οδηγία σε σχέση με την ε, προστασία ε, των καταγγελόντων και υπό την ιδιότητά μου αυτή απευθύνονται σε εσά. Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα στις 15 Ιουνίου και για πρώτη φορά είδαμε ότι τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κοινοβούλιο, το οποίο βρισκόταν, είχε ένα πρωτοπόρο ρόλο στην αφορά την πρόταση αυτή, αναγνωρίζεται ε, ένα νομοθετικό ευρωπαϊκό κείμενο, σε αυτό αναγνωρίζεται η ανάγκη να παρασχεθεί μια προστασία σε αυτούς που, οι οποίοι ε, οδηγούνται να αποκαλύψουν μια παρατυπία, μια παράνομη δραστηριότητα, μια επιλήψιμη πράξη και αυτό εις βάρος των, ε, της δικής τους επαγγελματικής ή προσωπικής ε, ζωής. Καταγγέλουν λοιπόν ε, κάποιο σφάλμα ή παρατυπία και πραγματικά τονίσαμε αυτή την ανάγκη. Η πρόσφατη επικαιρότητα του Lux της υπόθεσης των Panama Papers ε, μας έδειξαν πολύ καλά το ρόλο, τη σημασία και την χρησιμότητα ε, των ανθρώπων αυτών στην ε, ανείχνευση και την καταγγελία κάποιων πρακτικών μέσω των οποίων ορισμένοι παραβιάζουν, προδίδουν, παρακάμπτουν το γράμμα και το περιεχόμενο των βασικών, του νόμου και των βασικών μας αρχών. Ε, καταδικάστηκαν ε, δύο άτομα στο πλαίσιο της υπόθεσης ε, Lux Leaks και πολύ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την πεποίθηση ότι αν αυτή η ευηγία είχε εφαρμοστεί ε, στο Λουξεμβούργο τα πράγματα δεν είχαν πάρει αυτή την πορεία. Εν πάση περιπτώσει είναι ξεκάθαρο ότι τα σκάνδαλα δεν γνωρίζουν σύνορα η προστασία των καταγγελόντων θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο άρα η παγκόσμια προσέγγιση είναι απολύτω αναγκαία εδώ. Η κυρία Κοφεράτη έχει το λόγο. Ο κύριος Κοφεράτη, ευχαριστώ. Όπως ακούσατε, σας ζητάμε μια οριζόντια οδηγία για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους θαραλέους αυτούς ανθρώπους που αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους με μεγάλη ευθύνη που είναι πραγματικοί πολίτες της κοινωνίας και αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Χωρίς την εργασία αυτών των καταγγελόντων δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε τόσο έντονα και ζωηρά για τα θέματα αυτά φοροαποφυγής και φόρο φοροαπαλλαγής. που αφορούν πολλούς φυσικά πρόσωπα ή μεγάλες πολυεθνικές όπως δείχνουν και τα έγγραφα του Παναμά. Όπως ξέρετε και καταλαβαίνετε υποσκάπτουν τα θεμέλια της κοινωνίας μας και δυστυχώς αυτός που καταγγέλει τους υπεύθυνου δεν την χάνει προστασίας. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό το πλαίσιο. Νομίζω ότι για το κοινό μας συμφέρον οι άνθρωποι αυτοί, οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προστατεύονται από αυτή την οδηγία. Και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να τους προστατεύσουμε και τάχιστα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε, στο προσχέδιο ε, του κειμένου για τα εμπορικά μυστικά έχουμε δει ότι οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να μην ανακοινώνουν πληροφορίες τις οποίες πιστεύουν πως ε, πρέπει να διατηρηθούν εμπιστευτικές. Χρειαζόμαστε όμως κριτήρια για να στηρίξουμε αυτούς που καταγγέλνουν εκ των έσω, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε νομική ασφάλεια. Είναι σημαντικό να ε, λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να τους προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Σουρμπάν Κρέσπο, τα Panama Papers ε, κατέδειξαν ξανά την σημασία των καταγγελόντων για περιπτώσεις ε, φορολογικής ε, αποφυγής και άλλες περιπτώσεις διαφθοράς. Παρ' όλα αυτά αυτό που φαίνεται να ε, ε, απασχολεί τις ε, αρχές είναι το να, γίνει, να γίνουν απλώς γνωστά τα ονόματα. Η Κομισιόν υπέβαλε μια πρωτοβουλία για το εμπορικό, τα εμπορικά μυστικά τα, η οποία εκθέτει τους καταγγέλλοντες. Δηλαδή η Ντετούρ και η Αλέ τον καταδικάστηκαν ενώ οι καταγγελόμενοι ούτε καν δικάστηκαν είναι ε, η υπεράσπιση της δημοκρατίας σημαίνει υπεράσπιση του δικαιώματος της πληροφορίας και της αλήθειας. Ένα δικαίωμα για το οποίο οι καταγγέλλοντες κατα, ε, διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Υποχρέωσή μας είναι να τους προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε με βάση τις ε, επώνυμες καταγγελίες αλλά και τις ανώνυμες, το Κοινοβούλιο είναι ενωμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εάν και κατάφεραν οι καταγγέλλοντες να αποκαλύψουν σοβαρές υποθέσεις, δεν τα καταφέραμε να καταπολεμήσουμε την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή. Καμία κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς καταγγέλλοντες, είτε πρόκειται για, τον περιβάλλον, για το περιβάλλον, την οικονομία και τις κλιματικές αλλαγές. Θα πρέπει να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και γι' αυτό θα πρέπει να προβάλλουμε οριζόντια νομοθεσία για την προστασία των καταγγελόντων. Το ζητήσαμε, το ζητάμε εδώ και μήνες και το Συμβούλιο είναι έτοιμο να το προωθήσει. Γι' αυτό ακριβώς ε, μιλάμε για εποπτεία η οποία δεν αρχεί μετά από τους καταγγέλλοντες των LuxLeaks. Τι επιπλέον ε, αποδείξεις θέλουμε. Η Επιτροπή θα δεχτεί στο πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς να λάβει υπόψη την προστασία των καταγγελόντων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλή. Ευχαριστώ αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα με ξέπληξε, διότι δύο άνθρωποι που ήταν τίμοι και κατήγγυλαν τις σκανδαλώδεις πρακτικές της LuxLeaks, των LuxLeaks καταδικάστηκαν αντίστοιχα, αντίστοιχα σε ένα χρόνο και εννέα μήνες. Εμείς θεωρούμε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, της, ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Γιούνκερ, θα έπρεπε να δράσει. Ήταν πρωθυπουργό αυτή τη χώρα για 20 χρόνια. Τι έκανε, πού βρίσκεται η δικαιοσύνη εάν οι θεσμοί δεν κάνουν τίποτα και δεν προσπαθούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι οδηγούν την κοινωνία μπροστά. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη δραστηριότητα ε, ο κύριος Γιούνκερ την ε, συγκάλυψε για 20 χρόνια. Πιστεύω ότι οι δύο αυτοί καταγγέλλοντες ήταν πραγματικά ήρωες. Εμείς πιστεύουμε σε μια άλλη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο κ. Μάγερ δεν φαίνεται να είναι εδώ. Ο λόγος στην κυρία Ολσκου. Ε, Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή ε, που, την Προεδρία που ενήργησε τόσο γρήγορα εξ ονόματος της ομάδας των σοσιαλδημοκρατών μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι' αυτό γιατί είναι ιδιαίτερο ε, σημαντικό γιατί το να αποσιωπεί κανείς ε, το να προσπαθεί κανείς να φημώσει συγγνώμη, τους ανθρώπους που έχουν το κουράγιο να αποκαλύπτουν τις λειτουργίες, απάτες και παρατυπίες ε, δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να τους ανταμείβει κανείς και να τους προστατεύει μέσω του νόμου. Και η έκθεση που ψηφίστηκε σήμερα δείχνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει μάλλον να υποβάλει ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο το οποίο να εγγυάται την προστασία αυτών των ανθρώπων. Ε, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ε, χρειάζεται λοιπόν μια ε, υπήρξε μια ταχεία αντίδραση, αλλά χρειάζεται και μια υποβολή, ταχεία υποβολή μιας πρότασης επί της οποίας να μπορούμε να τοποθετήσουμε. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν ένα συγκεκριμένο απτό αποτέλεσμα, γιατί πρόκειται για μια σημαντική δυσλειτουργία και θα πρέπει να αντιδράσουμε τάχιστα. Ο κύριος Γκίγκολτ έχει το λόγο. Κύριε Κατάινεν, ε, απευθύνομαι άμεσα σε εσά. Γνωριζόμαστε από την εργασία στο πλαίσιο της ε, Νομισματικής ε, και Οικονομικής Ένωσης. Και θα έλεγα ότι για πέμπτη φορά σήμερα αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε επιτέλους ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελόντων. Ε, το ακούσαμε από όλε τι πολιτικές ομάδε από όλε τι πολιτικές αποχρώσεις. Οι πάντες επιθυμούν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ή να προτείνει μάλλον ένα οριζόντιο νομικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο είπε ότι ε, προτίθεται να το ακούσει. Ε, έκανε μια θετική κίνηση και θα ήθελα να ακούσω ξεκάθαρα από εσά. Πότε θα δείξετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να αναλάβει δράση. Πότε θα αποδείξετε ότι ο κύριος Γιούνκερ πραγματικά την ευήκον ους στο, στις προτάσεις του Κοινοβουλίου. Ε, αυτό το οποίο είπατε στη δική σας δήλωση δεν είναι επαρκές. Πότε, κύριε Κατάινεν, θα φτάσει ε, η πρόταση αυτή, ε, γιατί την αναμένουν με ανυπομονησία οι πολίτες της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρωσιέρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε το Swiss Leaks, LuxLeaks, τα Panama Papers. Ε, θα πρέπει να επικίνουμε και άλλο τη λίστα για να κρούσουμε το κόδωνα του κινδύνου. Ε, την περασμένη εβδομάδα ο Ραφαέλα Λέ και ο Αντουάν Ελτούρ καταδικάστηκαν από τη δικαιοσύνη του Λουξεμβούργου ενώ αποκάλυψαν το μεγαλύτερο σκάνδαλο οικονομικής απάτης ε, της δεκαετίας. Σήμερα ψηφίσαμε ε, τα πορίσματα του Tax 2 ε, για τα LuxLeaks. Ενώ η Ευρώπη διανύει μια κρίση χωρίς προηγούμενο, θα πρέπει να δείξουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι είμαστε σε θέση να δράσουμε στο όφελός τους και να προσπα... Ε, υπερασπίσουμε αυτούς που δρούν προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατικότητα. Αυτό το Κοινοβούλιο κάνει αυτή την συζήτηση σήμερα κατόπιν των σοσιαλδημοκρατών και αυτό το σώμα ζήτησε κατ' επανάληψη να υπάρξει μια τέτοια ευρωπαϊκή προστασία γιατί η προστασία σε εθνικό επίπεδο είναι ανεπαρκής. Θα πρέπει να, ενώ η απάτη είναι ευρωπαϊκής κλίμακας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια οριζόντια οδηγία έχουμε τα μέσα να βρούμε τη, μια βάση για να δράσουμε, να, προστασ... Ε, να παράσουμε μια προστασία με ένα οριζόντιο πλαίσιο. Ε, σας ζητώ λοιπόν κύριε Επίτροπε έχουμε, θα ήθελα να σας πω το εξής έχουμε ανάγκη μια πολιτική, μιας πολιτικής ε, βούλησης Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Τζαβόρ Αξιότιμε κύριε Επίτροπε αξιότιμοι συνάδελφοι κύριε Κατάενεν ο κύριος ε, Κατάινεν ε, μίλησε για κάποια μέτρα σε εθνικό επίπεδο. Εγώ πριν από μία εβδομάδα ήμουν στις, ε, στη δίκη του Αντουάν Λετούρ και το, η απόφαση η οποία λήφθηκε από το δικαστήριο είναι ξεκάθαρη έκφραση του γεγονότος ότι αυτό το οποίο είπατε ε, το οποίο δηλώσατε σήμερα δεν παρέχει επαρκή προστασία για τους καταγγέλλοντες. Δηλαδή οι παρόντες κανονισμοί και οι παρούσες οδηγίες δεν είναι επαρκείς ε, προκειμένου να υπάρξει μια αποτελεσματική προστασία των καταγγελόντων. Ε, δεν έχουμε πλέον άλλο χρόνο. Η καταδίκη του Λουξεμβούργου, του ε, αποστερεί από τις καταγγέλλοντες, ε, ε, τους απογεινώνει από το θάρρος, από την τόλμη την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Θα πρέπει να προστατεύσουμε επιτέλους αυτούς τους ανθρώπους και προκειμένου να προστατεύσουμε το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών πρέπει να γίνουν γρήγορα βήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κόφ. Επίτροπε, Εκπρόσωποι του Συμβουλίου. Μόλις, λίγες πριν από, ε, μόλις πριν από λίγες ώρες το Κοινοβούλιο με, με ισχυρότατη πλειοψηφία ε, ψήφισε ε, μέτρα προστασίας των ε, καταγγελών όπως ο κ. Σαλέο, κ. Περόν, ο Δελτούρ. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε διώξεις αυτών τέτοιων ατόμων. Επίσης δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το τι περιμένουμε από το Συμβούλιο και την Κομισιόν πλέον. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε ε, στι αρμοδιότητε των κρατών μελών, που δεν είναι. Όμω, αυτή τη στιγμή η ε, Ευρώπη ε, προδίδει τους καταγγέλλοντες ε, οι οποίοι έχουν το θάρρος και την παρουσία να καταγγείλουν τις παρατυπίες. Χρειαζόμαστε κύριε Επίτροπε ένα ισχυρό και συνεπές νομικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία τους. Χρειάζεται τα κράτη-μέλη να ε, δεσμευθούν σε ένα σύνολο ελάχιστων προδιαγραφών προστασίας ε, έτσι ώστε τέτοιου είδους καταγγελίες να γίνονται και στο μέλλον. Υπάρχουν πολλοί καταγγέλλοντε, που οι υποψήφοι καταγγέλλοντε που αυτή τη στιγμή φοβούνται τι διώξει. Είδαν τι έγινε στο Λουξεμβούργο. Πρέπει να σταματήσουμε την αυτόματη δίωξη των καταγγελόντων και να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να διώξουμε τους πραγματικούς εγκληματίες, όχι αυτούς τους ήρωες που καταγγέλουν, τους πραγματικούς υπέτειους των, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Συνεπώς, σας παρακαλώ πολύ, υποβάλλετε πρόταση σαφούς νομικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί τη χρειάζομαι τώρα, εδώ και τώρα. Αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η καταδίκη του καταγγέλλοντος Αντουάν Ντελτούρ είναι μια ήττα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να επαναληφθεί ποτέ. Δεν είναι δυνατόν ε, σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο να κινούμαστε με ρυθμό χελώνας προκειμένου να ε, καταπολεμήσουμε τη φορά αποφυγή και ταυτόχρονα καταδικάζουμε καταγγέλλοντες οι οποίοι ε, συνεισφέρουν κάτι εξαιρετικά πολύτιμο για την ε, δημοκρατία γιατί πρόκειται για μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δρούν παράνομα. Χρειαζόμαστε κατεπηγόντως στην Ευρώπη μια οριζόντια νομική ρύθμιση για την προστασία των κατακελώντων. Η Επιτροπή το τελευταίο διάστημα προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από νομικά επιχειρήματα λέγοντας ότι δεν είναι αρμόδια. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο κύριε Κατάινεν γιατί μια νομική, η νομική βάση υφίσταται. Άρα σας καλώ να την εφαρμόσετε. Η κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ πρόεδρε στον τομέα των αέριων μεταφορών, στον οποίο χρειαστεί πολύ, προστατεύονται απόλυτα αυτοί οι οποίοι καταγγέλουν παρατυπίες. Ε, εκεί το ονομάζουμε κουλτούρα της ασφάλειας. Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η ίδια κουλτούρα και για το δημόσιο συμφέρον. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται οριζόντια οδηγία προστασίας της ανωνυμίας των καταγγελόντων, θα τους δίδεται ε, νομική βοήθεια, συνδρομή και ψυχολογική συνδρομή ενδεχομένω. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως αυτές τις οποίες ανέφεραν συνάδελφοι, αλλά και άλλες πιο ανώνυμες περιπτώσεις, όπως στη χώρα μου, η Άννα Γαρίδο ε, και άλλοι που έχασαν τη δουλειά τους, χάλασε η ζωή τους, καταστράφηκε η ζωή τους επειδή ακριβώς για το δημόσιο συμφέρον κατήγγελαν παρατυπίες. Επίσης θα ήθελα να τιμήσω εδώ τον Μωυσές Βερμέχο της ΟΚΕ που μου έμαθε όλα αυτά τα πράγματα και ήταν ε, θύμα της ε, τόλμης του που ως υπάλληλο κατήγγειλε ε, διαφθορά εντός των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. η, η δίθεν ανυπαρξία νομικής ε, βάσης ε, άφησε έκθετο τον Μωυσές ε, τον οποίο θα ήθελα με αυτά τα λόγια να τιμήσω. Χρειαζόμαστε αυτή την προστασία και για τις μεγάλες και για τις μικρές υποθέσεις. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μαριάς έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε οι καταγγέλλοντες τις διάφορες παρανομίες δεν την χάνουν επαρκούς νομικής προστασίας στην ευρώπη. παρ' όλα αυτά οι καταγγελίες αυτές έχουν φανεί χρήσιμες στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. το σκάνδαλο luxleaks οι λίστες borgens και lagarde και φυσικά τα ονόματα επιφανών επιχειρηματιών και πολιτικών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας με τα panama papers κατέδειξαν ότι φυσικά πρόσωπα και πολυεθνικές επιχειρήσεις αποκομίζουν υπερκέρδη αποφεύγοντας να φορολογηθούν στα κράτη όπου λαμβάνουν χώρα οι δραστηριότητές τους. Και δυστυχώς κύριε Κατάινεν οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς γιατί μεταξύ άλλων κολλησιεργούν και οι ευρωπαϊκές αρχές. Τελευταία ήρθε να προσθεθεί σε αυτή τη λίστα και η αποκάλυψη για τις διαπραγματεύσεις της TTIP και η μυστική διπλωματία που ακολούθησε η Κομισιόν μετά τη διαρροή των απόρριτων εγγράφων η κομισιόν αναγκάστηκε να αλλάξει ρότα. η θέσπιση της προστασίας των καταγγελόντων που δρούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος είναι βέβαιο ότι θα αναδείξει και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις παραβιάσεων της νομιμότητας μέσα στην ευρωπαϊκή ένωση. είναι λοιπόν προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών να ενισχυθεί το πλαίσιο της προστασίας αυτών των ανθρώπων. ευχαριστώ. Όλοι μιλάμε για μεγάλα θέματα, έγγραφα του Παναμά, Λίξ, που είναι ευρέως γνωστά πλέον θέματα. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για αυτά, αλλά και για τους χιλιάδες καταγγέλλοντες που θέλουν να μας βοηθήσουν να καταπολεμήσουμε τα σκάνδαλα, τη διαφθορά τις παρανομίες των ε, μεγάλων επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να τύχουν προστασίας γιατί υπάρχει και διασυνοριακή διαφθορά και γι' αυτό χρειαζόμαστε όλο και περισσότερους καταγγέλλοντες. Στην Κροατία είχαμε μία γυναίκα καταγγέλουσα σε μία μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία η οποία ε, κατήγγειλε την επιχείρηση αλλά βρέθηκε σε μεγάλους μπελάδες. Το ίδιο ίσχυσε και με πληθώρα άλλων καταγγελιών. Ο κύριος Επιτίδιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαφθορά είναι μια παρεκτροπή η οποία είναι συμφασμένη με την ανθρώπινη φύση υπήρχε υπάρχει και δυστυχώς θα εξακολουθεί να υπάρχει σε όλα τα ηγετικά κλιμάκια των, ε, της διοικήσεως των επιχειρήσεων ε, των οργανισμών και των ε, πολυεθνικών σχηματισμών. ενώ όμως αυτό αποτελεί κοινό μυστικό και η διαφθορά βλάπτει πολλές φορές τα σφαίρα του κράτους είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν το θάρρος να καταγγείλουν πράξεις διαφθοράς και αυτό διότι ουδής προστατεύει. οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές γίνονται αντικείμενα διεκδικήσεως και ορισμένες φορές υφίστανται και ποινικέ διώξεις. αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο ηθικοί δεν είναι μόνο γενναίοι δεν είναι μόνο αξιέπαινοι είναι οι φύλακες του δημοσίου και του κοινωνικού συμφέροντος και αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να τους προστατεύουμε. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να θεσπίσει κανόνες προστασίας αυτών που αποκαλύπτουν τη διαφθορά διότι διαφορετικά γιατί να μην σκεφτεί κάποιο, ότι ο ηγετικό κύκλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το θάρρο να πολεμήσει τη διαφθορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατάινεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε από την ίδια πλευρά. Η, η πράξη αυτή είναι στοιχείο της ένομης τάξης στην Ευρώπη. Υποτίθεται θα πρέπει να είναι. Δυστυχώς δεν ισχύει κάτι τέτοιο σε όλες τις χώρες μέλη. Γι' αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να έχουμε μια στέρεη νομική βάση ούτως ώστε να προστατεύονται οι καταγγέλλοντες εφόσον προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας δώσω, να σας αναφέρω την, ε, ακριβή, την ακριβή ημερομηνία που θα υποβληθούν οι προτάσεις και θα πρέπει να αξιολογήσουμε το νομικό πλαίσιο. Ίσως αυτό σας φαίνεται κάπως βαρετό, αλλά ωστόσο όσον η προστασία των καταγγελών θα πρέπει να στηριχθεί στη νομική βάση και εμείς θα πρέπει να στηρίξουμε, να δρώσουμε τις προτάσεις μας σε ένα νομικό πλαίσιο. Ε, ορισμένες φορές θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποια είναι η αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ποια είναι η αρμοδιότητα των χωρών μελών. Ε, γνωρίζω ε, ε κατανοώ τα όσα λέτε για την αναγκαιότητα να υπάρξει μια επαρκή νομική προστασία στο πλαίσιο της ένομης τάξης και της δημοκρατικότητας. Ωστόσο η πραγματικότητα δεν είναι τόσο δεινή όσο ορισμένοι ε, θεωρούν εδώ. Παρόλο που υπάρχει βεβαίως ένα περιθώριο βελτιώσεων. Ε, υπάρχει μια νομική βάση την οποία ε, προβλέπουν οι συνθήκες αλλά πρέπει να κάνουμε μια σχετική αξιολόγηση. Οι διατάξεις αναφέρονται ε, σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος ε, και με, σε σχέση με την ε, πιστευτικότητα των εμπορικών δεδομένων αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει παρόλα αυτά να το αξιολογήσουμε και εμείς από την δική μας ε, πλευρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ισχυρή σας ε, πολιτική βούληση και εμείς από την πλευρά μας θα βρούμε τον ε, δρόμο να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα εκ μέρους του Συμβουλίου η κυρία Κορτσόκ, ο κύριος Κόρτσοκ, συγγνώμη. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση η οποία φώτισε το θέμα των καταγγελών των παρατυπίες και την προστασίας τους ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων ε, γεγονότων και υποθέσεων όπως υπογραμμίσατε πολλοί από εσάς. Όπως είπε και ο αντιπρόσκειος Κατάινεν πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η Κομισιόν αξιολογεί την ενδεχομένη ύπαρξη νομικής βάσης για την υποβολή πρότασης εγώ θα τελειώσω με τα αρχικά μου λόγια. Αν η Κομισιόν αναλάβει πρωτοβουλία, έχοντας ε, συμπεράνει ότι υφίσταται νομική βάση, τότε τον, ε, Ευρωπαϊκό, το Συμβούλιο θα ασχοληθεί με, με αυτή την πρόταση που θα υποβάλει η Κομισιόν. Όμως, παρόλα αυτά η συζήτηση ήταν ε, ιδιαίτερα σημαντική. Ωραία. Ολοκληρώνεται